Τα ψηφίσματα που επεγκρίθηκαν θα ε, διαβιβαστούν στα άτομα και τα ε, όργανα της φορείς που αναφέρονται σε αυτά τα ψηφίσματα. Πριν ολοκληρώσουμε, ε, σας